Uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε στη συνέχιση της χθεσινής μας συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Περνάμε στη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ιδίου σπόρους και του σχεδίου ανάκαμψης. Θα σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η διαπραγματεύσεις επιτέλους ξεκίνησαν με το Συμβούλιο για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και του ίδιου πόρου την περασμένη εβδομάδα. Ενώ, όπω ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ήδη έτοιμο για τι διαπραγματεύσει αυτέ εδώ και δύο χρόνια. Είχαμε ε, υιοθετήσει μια πολύ διεξοδική διαπραγματευτική εντολή για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και του ίδιου πόρου ήδη από τον Νοέμβριο του 2018. Βέβαια, η κατάσταση έκτοτε έχει εξελιχθεί και στεναρή εκείνη εντολή πρόσφατα τον Ιούλιο επικαιροποιήθηκε για να λάβει υπόψη και τη πρωτοφανή γεωνομική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες μας. Και από την πρώτη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι υπάρχει σημαντικό κενό, σημαντικό χάσμα μεταξύ των θέσεων του Συμβουλίου και των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει απτές βελτιώσεις στο πακέτο του Συμβουλίου. Και όχι μόνο δηλώσεις για να μας κάνουν ε, να μας βοηθήσουν να καταπιούμε το πικρό χάπι, όπως είπε και η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν. Γιατί η βασική μας ε, μέρημνα είναι να φροντίσουμε ώστε το επόμενο ΠΔΠ να είναι δεόντως εξοπλισμένο και για την ανάκαμψη αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των σημερινών μας εργασιών, θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στα πέντε μέλη της διαπραγματευτικής μας ομάδας για πέντε λεπτά στον καθένα. Μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις ηγητές για δύο λεπτά τον καθένα και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, μπορούν να λάβουν το λόγο. Πρώτα ο κύριος Γιάννη Όλμπριχτ από το ΕΛΚ που είναι και ο συνεισηγητής για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιάννη, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα αντικαθιστώ και την κυρία Μαργαρίτα Μάρκε τη συνεισηγήτριά μα, γιατί δυστυχώ απουσιάζει και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Οπότε θα μιλήσω και για τους δυο μας. Είμαστε συνεισηγητές για το τμήμα δαπανών του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου και τώρα περνάμε στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων είναι αρκετά περίπλοκη και ε, ασυνήθιστη, έκτακτη τελείως. Συνήθως, ε, για το πει, απαιτείται η συγκατάθεση, η συνένεση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο μετά τη λήψη των εγγράφων από το Συμβούλιο και είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη φορά όμως έχουμε την πρωτοφανή κατάσταση να έχουμε ένα ολόκληρο πακέτο. Ένα πακέτο από, την Επιτροπή πρώτα και από το Συμβούλιο και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ένα πακέτο που απαρτίζεται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο καταρχήν, από τον πολίτη, δηλαδή προϋπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζεται κυρίως σε εθνικές συνεισφορές και έχουμε και ένα επιπλέον προσωρινό μέσο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το Next Generation EU. Είναι το μέσο ανάκαμψης. Οπότε έχουμε ε, και το τρίτο στοιχείο, το κράτος δικαίου στο μέσο ανάκαμψης. Κάθε ένα από, τα, από τους μηχανισμούς αυτούς είναι διαφορετικός και διέπεται από διαφορετικές διαδικασίες. Ε, ο υποφαινόμενος και η κυρία Μάρκες ε, είμαστε αρμόδιοι, συναρμόδιοι για το ΠΔΠ, για το πρώτο σκέλος. Όπως είπε ο Πρόεδρος, έχουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του 2018 και επαναλαμβάνεται ή επιβεβαιώνεται με το τελευταίο μας ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι η μείωση των ε, βασικών δαπανών, δηλαδή των δαπανών για τις βασικές μας πολιτικές, που αφορούν ουσιαστικά τα εμβληματικά μας προγράμματα. Οι περικοπές αυτές ε, για τα εμβληματικά μας προγράμματα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να είχαν αντισταθμιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Μέσο Ανάκαμψης. Κάτι που δεν ισχύει όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γι' αυτό στο τελευταίο μας ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΠΔΠ και είπε ότι η τελευταία αυτή εκδοχή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου δεν είναι αποδεκτή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό σήμερα κρατούμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 15 βληματικά προγράμματα να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μεταξύ των προγραμμάτων αυτών δεν έχουμε την πολιτική συνοχή και την αγροτική πολιτική, γιατί αυτές δεν διακυβεύονται, τις προστατεύουν και τις υπερασπίζουν τα κράτη-μέρη. Τα εμβληματικά προγράμματα είναι το ορίζον, ο έρασμος, ε, ο έλεγχος των συνόρων, το Ταμείο Άμυνας και το καθεξής. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαριθμούμε αυτά τα 15 ευληματικά προγράμματα και τώρα ξεκινούμε τις διαπραγματεύσεις για τα προγράμματα αυτά και κυρίως για τα ανώτατα όρια, τις οροφές. Θέλουμε δηλαδή να πείσουμε το Συμβούλιο ότι αυτή η εκδοχή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι παράδεκτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί θα σήμαινε σημαντική μείωση των πολιτικών. Και για να συνοψίσουμε, ε, ισχύει κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται με τους οργανισμούς. Αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη των πολιτικών, θα πρέπει να μειωθούν οι πολιτικές και οι προτεραιότητες. Είναι σαφές. Και όταν συζητούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν συζητούμε χρήματα ουσιαστικά συζητούμε το πεδίο εφαρμογή και την εμβέλεια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν γίνουν δραστικέ περικοπέ στα κονδύλια των πολιτικών, εμεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε όχι μόνο στο Συμβούλιο αλλά και στου Ευρωπαίου πολίτε. «Συγγνώμη, λυπούμαστε πολύ, αλλά μην περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρηθούν αυτέ οι πολιτικέ, μια και το Ταμείο είναι μείον, δεν υπάρχουν κονδύλια για να τι χρηματοδοτήσουν». Οπότε ρόλο μα είναι να υπερασπίσουμε τη φιλοδοξία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη φάση λοιπόν έχουμε την εντολή και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με το Συμβούλιο τις δυνατότητες και τη μέθοδο για να ε, εξασφαλίσουμε αρκετά κονδύλια για πιο συγκεκριμένα εμβληματικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάν. Μια και απουσιάζει η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες η συνεισηγητρία, περνάμε στον ε, στον συνεισηγητή για το ΔΕΛΤΑΠ, τον κύριο Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα των ιδίων πόρων και για το θέμα των του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται με τους ρυθμούς, με φιλοδοξία και υπευθυνότητα. Σήμερα στην Επιτροπή Προπολογισμών θα υιοθετήσουμε την γνωμοδότησή μας για τους ιδίους πόρους και μάλιστα ε, δουλέψαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου για να διευκολύνουμε τις ε, συζητήσεις και να μπορέσουμε ήδη από τη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου να έχουμε την ψήφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με την ψήφο αυτή μπορούμε να περάσουμε στη διαδικασία της κύρωσης από τα κράτη-μέλη ανάλογα με τους συνταγματικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε ένωμη τάξη. Και ελπίζουμε την ίδια ταχύτητα να υιοθετήσει και το Συμβούλιο. Και θα πρέπει και το Συμβούλιο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Γιατί χωρίς την κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη, ανάλογα, όπως σας είπαμε, τους συνταγματικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος, δεν ε, θα έχουμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και αυτό το πακέτο ε, περιλαμβάνει και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο ανάκαμψης ή το Ταμείο Ανάκαμψης η απόφαση για τους ιδίους πόρους είναι ιστορική. Για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια έχουμε και νέο ιδιοπόρο, το φόρο για τα πλαστικά. Και επίσης δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα να δανειστεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να μετατρέψει αυτά τα δάνεια ε, σε ε, επιδοτήσεις. 390 δισεκατομμύρια θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε μετά το 2021 τους πολίτες, ούτε να κόψουμε το ε, ΠΔΠ μετά το 2027. Γι' αυτό λέμε ότι μετά το 2021 θα χρειαστούμε νέους ίδιους πόρους. Με βάση την απλούστατη αρχή, όποιος δεν πληρώνει θα πρέπει να πληρώσει. Οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βοηθήσουν για να καταπολεμήσουμε και τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους και για αυτές τις αρχές, προτείνουμε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για, τη, για τους ίδιους πόρους που θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι από το 2021 και θα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκής για να αποπληρώνουμε τα επιτό... τους στόκους και τις αποσβέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το Next Generation EU, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών, κανένας δεν αντιλαμβάνεται πώς είναι δυνατόν το ταμείο αυτό να μπαίνει στον προϋπολογισμό χωρίς να έχει λόγο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Θέλουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, γιατί μερικές φορές πρέπει να υπερασπίζουμε και το Συμβούλιο με τα λεγόμενά μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι δύο βραχίονες της ε, Δημοσιονομικής Αρχής να έχουν μια αιτήσια διαδικασία ώστε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να ακολουθούν τις γραμμές και τις προτεραιότητες στις οποίες θα συμφωνήσουμε. Και είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Είναι θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, ε, σαφήνειας, διαφάνειας, λογιστικού ελέγχου. Θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους την χάνουν αξιοποίησης με διαφάνεια. Γι' αυτό αλλάζουμε το δημοσιονομικό κανονισμό, γι' αυτό αλλάζουμε και τη διοργανική συμφωνία και έχουμε τη λύση για να εξασφαλίσουμε αυτή τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και ας μην ξεχνούμε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μυαλό μας είναι 750 δισεκατομμύρια ευρώ. 360 ε, για δάνεια και 390 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις. Εμείς θέλουμε όλα αυτά τα χρήματα να πιάσουν τόπο, να χρησιμοποιηθούν με χρηστό τρόπο και να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο. Επίσης, αν τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιηθούν, δεν απορροφηθούν, θα θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα επαναφέρουμε στο υπεροπολογισμό για τα εμβληματικά προγράμματα που μας ανέφερα ο προλαλής σας. Και αυτός είναι ένας στόχος που ελπίζω να εστερνιστούν και όλα τα κράτη-μέλη, όπως πιστεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Ζωζέ Μανουέλ. Και τώρα η κυρία Αγέρ από την Ρινιού και εκείνη συντονίστρια για το θέμα των ιδίων πόρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το θέμα των ιδίων πόρων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας αγώνας που δίνουμε όλοι μαζί από καιρό κρίση και η απάντηση που δόθηκε στις ανάγκες μας με αυτόν τον προπολογισμό, αυτά που έχουμε προτείνει και εμείς ως Ευρωβουλευτές, δίνουν επιπλέον επιχείρημα στο Κοινοβούλιο για να προχωρήσει και να συνεχίσει να πιέζει για το θέμα των ίδιων τρόπων. Η απάντηση του Συμβουλίου, αν και αρχική κρατών και κυβερνήσεων αποφάνθηκε για το θέμα ε, στα συμπεράσματα της 21ης Ιουλίου, ε, περιλαμβάνουν, έχουν περιλάβει πολλά στοιχεία που δεν μας ικανοποιούν. Η αρχή της δανειδότησης και επιστροφής ε, δανείων από τους ίδιους πόρους ήταν κάτι που καθορίστηκε. Ωστόσο, και εκεί φαίνονται οι αδυναμίες της συμφωνίας, τα συμπεράσματα ε, αφήνουν ένα παραθυράκι για κάποια κρατημέλη. Γιατί το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται δεν είναι αρκετά δεσμευτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 θα πρέπει να επιβάλλει, φόρο, θα πρέπει να επιβάλλει προτάσεις για τη φορολόγηση των μεγάλων ψηφιακών εταιριών και την ε, πρόβλεψη νέων δασμών. Εδώ θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να πιέσουμε για νέους ιδίους πόρους. Ε, πρέπει να δούμε και αν ε, το ε, σύστημα ανταλλαγής εκπομπών θα είναι μια πηγή για τους ίδιους πόρους. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν αφήσει και άλλα παρατηράκια στο παρελθόν, όπως κάνουν και τώρα, και εδώ και 32 χρόνια ζητάμε μεταρρύθμιση του συστήματος ίδιων πόρων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ δεν αναφέρεται καν πώς θα γίνεται η επιστροφή των ε, ποσών από το σύστημα των ίδιων πόρων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να συμφιλειώσουμε το πνεύμα της συζήτηση με τα κείμενα που υιοθετούνται. Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα δεσμευτικό, ώστε και τα δύο μέρη των διαπραγματεύσεων να μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ένα χρονοδιάγραμμα ε, κάπως πιο γοργό Πράγμα που θα δούμε και στην γνωμοδότηση που θα εγκρίνουμε σήμερα το απόγευμα. Και θα πρέπει να υπάρχει μια διαθεσμική συμφωνία ώστε να αποφύγουμε κάθε είδου κλειδονισμού στο μέλλον και να έχουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων που να εγκριθεί πλέον μια και καλή. Ε, θα πρέπει να κλείσω εδώ λέγοντα ότι ο αγώνα αυτό είναι ζωτική σημασία γιατί όπω είπε ο Ζωζέ Μανουέλ προηγουμένω υπάρχουν τρει επιλογέ για να επιστραφούν τα δάνεια. Οι νέοι ήδη πόροι ή η περικοπή των προγραμμάτων ε, συνολικά στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου ε, ή κάτι άλλο. Και βεβαίως εδώ εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών δεν θέλουμε ε, να μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις που υποφελούνται από τις ευνοϊκές συμφωνίες, τις φορολογικές συμφωνίες και θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτέ στην ανοικοδόμηση. Και ακόμη μερικά σχόλια. Έχω λίγο χρόνο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω καταναλώσει ήδη. Ε, ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ο προπολογισμό αυτό είναι πραγματικά θέμα αριθμών, αλλά όχι μόνο. Είναι και θέμα πολιτικών ε, φιλοδοξιών. Εδώ πρέπει να πω ότι η επιστολή των τεσσάρων πολιτικών ομάδων, ΕΛΚ, ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ρινιού και Πρασίνων, αναφέρει ότι η κατάσταση στην Ευρώπη τώρα μας ε, αναγκάζει να αναλάβουμε δράση ε, και λόγω της, ε, των περιορισμών των ελευθεριών των πολιτών, της ελευθερία του τύπου, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια αγορά, είναι και μια κοινότητα αξιών. Αυτό ισχύει και οι αξίε αυτέ έχουν εγκριθεί από τέτοια τα κράτη-μέλη όταν ενέκριναν ε, και ψήφισαν τι συνθήκε μα. Αυτό λοιπόν ζητούμε, να γίνουν σεβαστέ οι αρχέ και οι συνθήκε που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν. Δεν τα λέμε αυτά για να εξοραίσουμε την κατάσταση, δεν είναι μια άσκηση καλοπιστική, αλλά θα πρέπει να βρούμε αυτού του ζωτικού μηχανισμού που θα μα επιτρέψουν ε, να ε, σχηματίσουμε τέτοιου συναρπισμού ώστε στην πραγματικότητα να βρούμε λύσει. Ευχαριστούμε, Βαλερή. Τελευταίο από τη θυμοτευτική ομάδα, ο Ράσμου Άντρεσεν από του Πρασίνου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω τρεις ε, παρατηρήσεις σε αυτά που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, τους οποίους υποστηρίζω εν γέννη. Νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη, όπου κάποια από τα θέματα είναι πιο περιπεπλεγμένα από άλλα, όπως το κράτος δικαίου. Θέμα εξαιρετικά περίπλοκο και φαίνεται τώρα ότι ανακύπτει το ζήτημα των επιμέρους προγραμμάτων. Θα είναι και αυτά πολύ περίπλοκα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αποστείλουμε κάποιο ισχυρό μήνυμα για τα επιμέρους προγράμματα όπως είπε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Όλμπριχτ, Είχαμε συγκεκριμένε επιταγέ για το τι πρέπει να κάνουμε και αργότερα στο Γερμανό Υπουργό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι αποδεκτό να έχουμε διπλωμάτες και να κυκλοφορούν διπλωμάτες που λένε ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να αποδεχτεί το ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσει στα ε, χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών, γιατί λιγμών άλλω ήταν πολύ δυσχερή η διαπραγματεύση στο Συμβούλιο, κράτησαν πάρα πολύ και θα πρέπει το Κοινοβούλιο αναγκαστικά να αποδεχτεί το πόρισμα του Συμβουλίου. Εδώ πρέπει να ε, ανακοινώσουμε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό για το Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να έχουμε σκληρή ε, διαπραγμάτευση για το θέμα των επιμέρους προγραμμάτων και νομίζω ότι τουλάχιστον η Γερμανική Προεδρία θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν θέλουν, για παράδειγμα, αύξηση στον προπολογισμό του προγράμματος για την υγεία ή τα άλλα προγράμματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Αυτά βλέπω εγώ σε σχέση με το που βρισκόμαστε ε, ως προς τα επιμέρους προγράμματα τώρα. Πάντως θα πρέπει να συζητήσουμε και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, να επιμείνουμε για τα οριζόντα διαθέματα, όπως την ενδιάμεση αναθεώρηση, ε, αλλά και το θέμα του κλίματος. Ε, εδώ χθες Συζητήσαμε το θέμα της μελέτης για το κλίμα και είδαμε εκεί να υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τους μηχανισμούς. Τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο που παρακολουθούμε και χνηλατούμε από τη σκοπιά του κλίματος το τι συμβαίνει με τα βιοπικιλότητα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς μηχανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώ μεταβάλλει το πώς ε, μετρά ποσοτικά τα θέματα του κλίματος, το, τη διάσταση τη βιοπικιλότητα. Το ίδιο και για το φύλλο. Η συνάδελφος η κυρία Μάρκες μου είπε ότι το 1990 ε, εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε ασχολείται ήδη με τα θέματα του φύλου και ε, ήδη από τότε δεν ήταν ξεκάθαρο το τι κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε με την Γερμανική Προεδρία ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καθορίσουμε κάτι σαφές. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικότερο που θα πρέπει να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο είναι ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε ενιαίο μέτωπο. Και να φανεί ότι έχουμε την ίδια ευρεία πλειοψηφία που έχουμε και του προηγούμενου μήνε. Εάν δεν γίνει αυτό, θα αποδυναμωθούμε. Και κανεί από εμά δεν θα καταφέρει να προωθήσει τι προτεραιότητε που έχει ενδεχομένω η κάθε πολιτική ομάδα ξεχωριστά. Αυτό είναι ε, άκρο σημαντικό. Όχι για να αγχωθούμε, αλλά για να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και ότι μπορούμε να αγωνιστούμε και να διαπραγματευτούμε σκληρά με την διάθεση να επιτύχουμε κάποια συμφωνία εν τέλει και όχι να εμποδίσουμε κάποια συμφωνία, αλλά να έχουμε πραγματικά ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Ε, το είπαμε όλοι οι συνάδελφοι και στην προηγούμενη Σύνοδο Ολομέλειας. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Το επιχείρημα της πίεσης χρόνου που ήδη χρησιμοποιούν κάποιοι σε δημόσιες εκδηλώσεις κατά το Κοινοβουλίο είναι ένα επιχείρημα κακό, διότι το Συμβούλιο πρότεινε την ε, λύση που πρότεινε, εμείς είμαστε έτοιμοι, ήδη από αυτή τη συνάντηση φαίνεται ότι θέλουμε να συζητήσουμε. Το Συμβούλιο δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα του, της έλλειψης χρόνου. Περιμέναμε δύο χρόνια για να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Είναι πολύ καιρό. Εάν υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποια προγράμματα, δεν θα φταίει το Κοινοβούλιο θα φταίει το Συμβούλιο με τη στάση του και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ευχαριστούμε, Ράσμους. Να δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις ε, εισηγητές για δύο λεπτά ο καθένας. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κόρναν από τους Ρινιού. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα εδώ και κάθε φορά που η διαπραγματευτική μας ομάδα μας παρουσιάζει ε, τις προτεραιότητες εδώ και τα όσα έχουν συζητηθεί, ε, το θίγουμε ξανά και ξανά, αλλά τώρα νομίζω πως έχουν προχωρήσει τα πράγματα, δηλαδή έχει φτάσει πλέον η χρονική στιγμή όπου πρέπει να κάνουμε κάτι, έχουμε και τη Γερμανική Προεδρία ε, του Συμβουλίου, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι ουσιαστικά να παραμερίσουν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους ζητήματα, γιατί έχουμε ε, συζητήσει τα ε, επιμέρους ζητήματα στα διάφορα ψηφίσματά μας. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο τι θα πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν εγώ δημοσίω, για παράδειγμα και με τον τύπο, συζητώ τις προτεραιότητες ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω την αίσθηση ότι η κοινή γνώμη βρίσκεται ε, στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κυριότερα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και επίση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει πολίτης που να θεωρεί ότι δεν πρέπει να λάβουμε κάθε μέτρο προκειμένου να ε, προστατέψουμε το ε, κράτος δικαίου. Από εκεί και μετά όμως αυτό που μας λένε οι δημοσιογράφοι είναι ότι εσείς ως κοινοβούλιο δεν θα καταφέρετε να επιβληθείτε έναντι του Συμβουλίου. Και εκείνο που απαντάω εγώ είναι το εξής. Ε, το, κοινοβούλιο αυτό εδώ ε, είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια και όπου ήταν ε, διασπασμένο αν θέλετε. Νομίζω πως δείχνουμε τώρα ένα κοινό μέτωπο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη συνοχή. Και από εκεί και μετά θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να επιμείνουν σε αυτό προκειμένου ακριβώ να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια κοινή ενιαία στάση, να υπάρξει και συνοχή μεταξύ μα. Οπότε σε κάθε βήμα της διαπραγματευτική διαδικασίας θα πρέπει να καθιστούμε πολύ σαφή τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να την εκφράζουμε προς τα έξω. Και από εκεί και μετά ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κράτου δικαίου θα πρέπει να επιμείνουμε. Δηλαδή, εάν μέσα σε αυτό το ε, ε, επόμενο πακέτο, με το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν εντάξουμε και τι αιρεσιμότητε σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, νομίζω πω θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε στο μέλλον. Και πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σημαντικό αφού θίγει τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Οπότε α συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων από τη δική μα πλευρά, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Και νομίζω πω αυτέ τι πιέσει τι ασκεί με πολύ επιτυχημένο τρόπο η διαπραγματευτική ομάδα, ε, την οποία την ευχαριστώ για αυτό αυτό και νομίζω πως ε, ε, σήμερα θα θέσουμε και ένα πολύ ξεκάθαρο ε, ζήτημα και θα ταχθούμε και θα θέσουμε πολύ ξεκάθαρα τη θέση μας απέναντι στο Συμβούλιο ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε απέναντι σε πιέσεις που θα μας ασκηθούν. Ευχαριστώ, Λέω ο Πρόεδρος, ο κύριος Ζανιάντη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν άκουσα το πρώτο κομμάτι της συζήτηση ε, που κάναμε, αλλά όπως γνωρίζετε δεν είναι εύκολο τη σήμερα ημέρα να καταφτάσει κανείς στις ε, Βρυξέλλες ε, με αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, έχω παρακολουθήσει το όλο ζήτημα, έχω παρακολουθήσει τις, τη δουλειά που έχει γίνει και από την πλευρά της διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά και από την πλευρά της ομάδας επαφής ε, του Σασόλου. Οπότε γνωρίζω πως γίνονται κάθε προσπάθειες από τη, κάθε προσπάθεια από τη δική μας πλευρά και αντιμετωπίζουμε πιέσεις. Και εγώ λοιπόν από την πλευρά μου θα ήθελα να θέσω ε, δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι ε, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινοβούλιο, περισσότεροι τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, το επόμενο πακέτο, είναι το κράτος δικαίου ειδικότερα και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν κάποια από την πλευρά του Συμβουλίου τα οποία έχουν ταχθεί κατηγορηματικά κατά αυτής της λύσης και με αυτόν τον τρόπο βέβαια είχαμε ένα ζήτημα και σε ό,τι αφορά και το, ε, τη συμφωνία ανάκαμψης, αλλά από εκεί και μετά έχουμε και το δεύτερο ζήτημα των ιδίων πόρων που μας απασχολεί. Εδώ λοιπόν, εάν θέλουμε η ε, να είναι λίγο πιο ευρία η λύση την οποία θα βρούμε σε ό,τι αφορά τους ε, δύο σπόρους, τότε θα πρέπει ε, να υπενθυμίσουμε και στα κράτη-μέλη ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί ή να είχε επιδιωχθεί ήδη και τότε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, του Ιουλίου. Οπότε νομίζω πως η προτιμητέα στρατηγική για μας και πολύ πιο χρήσιμο, πολύ πιο χρήσιμο, θα ήταν να εστιάσουμε σε πολύ συγκεκριμένα ε, στοιχεία του υπροπολογισμού και να τα ε, θέσουμε εκ νέου επιτάπητο ε, εφόσον υπάρξουν εκεί περικοπέ. Αναφέρομαι εδώ για παράδειγμα στην κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει εδώ νομίζω συμφωνία ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. Και παρότι έχουν προσθεθεί νέε προτεραιότητε, εξακολουθεί να αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο διέρχεται μια δύσκολη περίοδο και γι' αυτό θα πρέπει να λάβει υποστήριξη. Και εδώ αναφέρομαι βέβαια και στι πιέσει που δέχεται σε παγκόσμιο επίπεδο και στι αλλαγέ οι οποίε λαμβάνουν χώρα σε ό,τι αφορά ε, τι εφοδιαστικέ αλυσίδε στο επίπεδο τη παραγωγή τροφίμων. Οπότε εδώ νομίζω πω θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουμε συγκεκριμένα σε αυτή την πολιτική για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Να έχουμε δηλαδή με φιλοδοξία εδώ, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα ρεαλιστικοί. έχοντα ε, πάντα κατά νου ε, τα δύο αυτά πιο ε, δύσκολα ζητήματα του κράτους δικαίου και των ιδίων πόρων. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επιμείνουμε τόσο, για παράδειγμα, σε τοπικά ζητήματα όπως αυτό των ιδίων πόρων, όταν έχουμε άλλα πιο σημαντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η περικοπή κονδυλίων που είναι εξαιρετικά ε, ανησυχητικό. Ο κύριος ε, Ζήλε τώρα από το ECR, λέει ο πρόεδρος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που αναφέρθηκε ότι δηλαδή ότι έχουμε μια ανάμειξη εδώ του νέου μέσου ανάκαμψη με το του δημοσιονομικό πλαίσιο και τα παραδοσιακά μέσα. Αυτό λοιπόν που είπε ο Γιάννα Αρμπίχτη, ότι αυτή, αυτή η μίξη που γίνεται είναι κάπω προβληματική θα πρέπει πραγματικά να δούμε ε, σε βάθος χρόνου τι, τι, τι έχει γίνει και από εκεί και μετά ε, είναι αυτό και αυτό που υπόθηκε σε ό,τι αφορά το, το, το επιχείρημα εκείνο ότι βρισκόμαστε υπό, υπό πίεση ε, χρόνου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ε, συμβαίνει είναι ότι το Συμβούλιο δεν πρόκειται να διασπάσει αυτό το πακέτο και από εκεί και μετά υπάρχουν και ε, πιέσεις που ασκούνται από εκείνους οι οποίοι ενδεχομένω θα είναι δικαιούχοι αυτό το κονδυλίο του, του, του, του μέσου ανάκαμψης. Βέβαια, ε, σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε, η ανάκαμψη, η ίδια διαδικασία της ανάπτυξης έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα όπως στη Γερμανία, ε, χωρίς να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέσου ανάκαμψης. Αντιθέτως, σε σε χώρες, για παράδειγμα του Νότου, τα πράγματα είναι δυσκολότερα και εκεί ενδεχομένως αυτό το επιχείρημα της χρονικής πίεσης να είναι και πιο σημαντικό. σε ό,τι αφορά τώρα ε, το μηχανισμό ανάποκριση να πούμε ότι ε, προφανώ υπάρχει εδώ μια διαφοροποίηση γιατί το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ε, βασίζεται σε εθνικού φακέλου, ε, στα, εθνικά κομμάτια, αν θέλετε, τα κονδύλια ενώ έχουμε από εκεί και μετά άλλα ε, κομμάτια, για παράδειγμα όπως ε, το Connecting Europe Facility, ε, άλλα στοιχεία όπως το Erasmus και άλλες, άλλες πολιτικές συνδικότητες, ή το Horizon για παράδειγμα, που έχουν διαφορετική φύση και έχουν ένα πιο κοινό χαρακτήρα. εμείς από την πλευρά ε, του ECR ε, θα μπορούσαμε να ε, συμφωνήσουμε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα. Θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο οδικό χάρτη σε ό,τι αφορά δηλαδή τους ιδίους πόρους. Ε, και το πώ ακριβώ αυτή θα εξασφαλίζεται και όχι δηλαδή με μείωση αυτών των ιδίων πόρων μέσα στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, Κάποιο ανέφερε ότι οι ε, ε, πολίτε των τρίτων χωρών θα κληθούν τελικά να, να επομιστούν, αν θέλετε, την επιβάρυνση που θα προκύψει από την αναδιάθρωση αυτών των ιδίων πόρων. Ε, εντάξει, φυσικά όταν υπάρχουν αλλαγέ σε πολιτική, καλούνται οι καταναλωτέ να υπομισθούν αυτό το βάρο ή άλλοι δικοί μα ε, πολίτε. Οπότε νομίζω πω αυτό δεν αποτελεί έγκυρο ε, πολιτικό επιχείρημα. Ε, δηλαδή, για ένα δικό μα μηχανισμό, ένα δικό μας οικονομικό εργαλείο των επιβαρυνθούν πολίτες τρίτων χωρών δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που μας απασχολεί με, αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος βλέπω κάποιες χειρονομίες εδώ, κάποιον εκνευρισμό, οπότε ε, να πω ότι ακούμε καταρχήν εδώ τους σκιώδεις εισηγητές, δηλαδή ακούσαμε τους Κέρνερ, Ζάνη και Ζήλε και θα ακούσουμε συνέχεια τον κύριο ε, Παπαδημούλη και συνέχεια θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ιδίων πόρων. Έτσι έχουμε διαρθρώσει τη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημούλης έχει τώρα το λόγο, αλλά δεν, ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, οπότε ο κύριος Κόκαλης θα διαβάσει το μήνυμα που έχει προετοιμάσει ο κύριος Παπαδημούλης. Παρακαλώ. President. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρει λοιπόν ο κ. Παπαδημούλη ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για να χάσουμε στι διαπραγματεύσει μα. Ε, ε, συγχαίρω την διαπραγματευτική ομάδα, ε, γιατί βέβαια ο ιό έχει επανέλθει, συνεχίζει να μα ασκεί πιέση και να αποδυναμώνει τι οικονομίε μα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια χρονική συγκυρία που αντιμετωπίζουμε την σημαντικότερη κρίση τη δική μα γενιά, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των μελλοντικών γενιών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια από τη δική μα πλευρά, από κοινού με την αρχή προπολογισμού, προκειμένου να επανέλθουμε ε, ισχυρότερη και με ανθεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, βοηθήσουμε τους πολίτες στις προκλήσεις που αντιμετωπίσουν και πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε περισσότερο την βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Ωστόσο, ε, τα κονδύλια τα οποία έχουν προβλεφθεί για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν επαρκούν ε, για την επίτευξη των πολιτικών που έχουμε αναφέρει. Ε, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το 30% των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί για την Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, θα θέλαμε να δούμε πώ θα διαμορφωθούν και πώ θα κατανεμηθούν. Και βέβαια δεν επαρκούν με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε του στόχου που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρεσίων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει περισσότερη προσπάθεια και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν θα ευθυγραμμίζεται ε, πλήρως με την ε, ε, Συμφωνία των Παρισίων και θα βασίζεται σε επιστήμες. Και επίση θα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία που έχει προταθεί από το Συμβούλιο τη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε εδώ ότι η τελευταία μεταρρύθμιση του συστήματο των ιδίων πόρων έλαβε χώρα πριν από 32 χρόνια. Οπότε ε, η δική μα στάση είναι ότι σε κάθε περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εγκρίνει το επόμενο ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο χωρί να συνοδευτεί και από αυτή τη νέα πρόταση για του ίδιου πόρου. Χρειαζόμαστε μια άμεση δεσμευτική πρόταση για του ιδίου ε, πόρου η οποία να καλύπτει με τον αποτελεσματικό τρόπο το, το κόστος για τα επόμενα προγράμματα, τον προπολογισμό και επόμενα προγράμματα και προκειμένου να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, για παράδειγμα όπω ε, και την ε, εκτριακή βιωσιμότητα ε, και χωρί να υπάρξουν αρνητικέ επιπτώσει σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόκαλη που αντικαταστήσατε τον κύριο Παπαδημούλη. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις συγητές για τους ιδίους πόρους. Η κυρία Κουαλμίνη από τους Έλληνε Δημοκράτες πρώτα. Ε, Δυστυχώς έχουμε μόνο ήχο και ο ήχος δεν μεταφράζεται. If we don't see you, uh, you... από τη στιγμή που έχουμε μόνο ήχο και όχι εικόνα, δεν πρόκειται να σας ε, μεταφράσουν οι τερμινείς. Αν θέλετε να μεταφραστείτε, παρακαλώ, ανάψτε και την κάμερά σας για να έχουμε και εικόνα.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 σας ευχαριστούμε κυρία Γκολμίνη. Η κυρία Λαπόχτ τώρα έχει το λόγο από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τους ιδίους πόρους, ε, 755 δισεκατομμύρια θα δανείσει στις αγορές Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 390 δισεκατομμύρια θα δώσει επιχορηγήσεις και 360 σε δάνεια. 1,514 είναι το ΠΔΠ. Ε, επίσης, ένα μεγάλο κονδύλι θα πάει στα πιο πληγέντα κράτη και μάλιστα θα επιχορηγηθεί όχι από τους δικαιούχους, αλλά από το σύνολο των Ευρωπαίων. Θα έχουμε δηλαδή μια μεταφορά χρημάτων μέσω ενό κοινού δανεισμού. Πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αποπληρώσει αυτό το νέο δάνειο που θα συνάψει. Μα λένε ότι οι, Ευρω... οι αμερικανικέ ή οι κινέζικε επιχειρήσει δεν ε, επίση λαμβάνουν επιχορηγήσει. Γιατί δεν σκεφτήκαμε εμεί νωρίτερα κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρο μα, ο κύριο Μακρό, μα εξήγησαν ότι ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Ευρωπαίοι γενικώ δεν θα χρηματοδοτήσουν αυτέ τι επιχορηγήσει. Αν όμως ε, έχουμε ψηφιακό φόρο, το φόρο προσαρμογή στον άνθρακα και στα πλαστικά που θα πλήξουν τι μεγάλε πολυεθνικέ, τι θα γίνει αντικειμενικά και σε τελική ανάλυση. Σε ποια ε, ταμεία θα μπουν αυτά τα κονδύλια στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές με τους ίδιους πόρους. Ε, βέβαια, οι επιχειρήσεις έχουν πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά έξοδα και δαπάνες. Και τι θα γίνει με τα επιδόματα ανεργίας. Μήπως τελικά ε, οι, επιχορηγήσεις, ε, ε επιχειρήσεις θα αυξήσουν τα προϊόντα τους και έτσι σε τελική ανάλυση συγκαλυμμένα θα πληρώσουν τα σπασμένα τα νοικοκυριά που θα πρέπει να αγοράζουν πιο ακριβά προϊόντα. Τίποτα δεν μας εγγυάται ότι οι νέοι διπόροι εκτός από το φόρο για τα πλαστικά που θα ισχύσει από του χρόνου, ότι θα θα εφαρμοστούν από το 2027. Ε, για τα φορολογικά θέματα απαιτείται ομοφωνία των ε, κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό φόρο στις μεγάλες πολυεθνικές, δεν φαντάζομαι η Ιρλανδία να δώσει το πράσινο φως για ένα τέτοιο φόρο στους ε, κολοσσούς ε, του ψηφιακού κλάδου. Τελικά κάθε μήνα, κάθε χώρα θα πρέπει να δίνει τη συνεισφορά της, εκτός και αν γίνουν πολύ σημαντικές περικοπές ε, ε, στα προγράμματα μέχρι το 2035. Πρόκειται να, να τροποποιηθεί η ομοφωνία στα φορολογικά και να περάσουμε στην ενισχυμένη πλειοψηφία. Επίσης, αν οι ήδη πόροι δεν υλοποιηθούν μέχρι το 2023, ποια θα είναι η εναλλακτική που προτείνετε. Ευχαριστώ κύριε Λαπόρτ. Ο κύριος Κόρμαντ έχει το λόγο από τους πράσινους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε ε, ένα μετέχνιο της συζήτησης, αλλά και σε ένα νευραλγικό σημείο ε, για το μέλλον της Ευρώπης και για την ιδέα που θα έχουμε για το μέλλον αυτό. Από τα θέματα που συζητήσαμε, είναι σημαντικό το θέμα της ε, κυριαρχίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι το δημοκρατικό όργανο και θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για τις δαπάνες. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το θέμα των ιδίων πόρων αντιλαμβανόμαστε αυτό τον εκβιασμό και μετράω τα λόγια μου, τον εκβιασμό που κάνει το Συμβούλιο εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας λέει ότι θα πρέπει να υποχωρήσετε στο ΠΔΠ, στους ίδιους πόρους και στη δημοκρατική σας κυριαρχία να αποφασίσετε για τις δαπάνες λόγω του, της υγειονομικής έκτακτης ανάγκης και ότι θα πρέπει πάση θυσία να υποχωρήσουμε, να ενδώσουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάγκη. Ή θα ε, δεχτούμε λοιπόν να εσωτερικεύσουμε αυτόν τον εκβιασμό, είτε θα θεωρήσουμε ότι αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική για να ανακτήσουμε τη δημοκρατική μας κυριαρχία. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε. Και αυτό θα είναι και το μέσο για την μελλοντική αλληλεγγύη. Θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο. Δικαίω πολλές χώρες υποφελήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη με το μέσω ανάκαμψης. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οι ίδιοι πόροι του σήμερα θα εξαρτήσουν την αυριανή αλληλεγγύη. Και αν δεχτούμε αυτούς τους ίδιους πόρους, που είναι δίκαιοι οι ίδιοι πόροι, δεν μιλούμε για δίκαιη φορολογία, ε, μιλούμε για όσους σήμερα φοροαποφεύγουν και αυτοί θα πρέπει να φορολογηθούν. Και πιστεύω ότι αν έχουμε την κρίσιμη μάζα και τη συγκεντρώσουμε, θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτά τα χρήματα για να έχουμε μια ουσιαστική αλληλεγγύη. Θα ήθελα λοιπόν να εφαρμόσουμε μια πυγμή, ήρεμη πυγμή και αποφασιστικότητα, την ηρεμία των παλέμαχων σε αυτή την ιστορική στιγμή, αλλά να δείξουμε μια αμήλικτη αποφασιστικότητα. Ε, έκανα, έχουμε μια πρόταση την οποία ψηφίσαμε. Εμεί τη δουλειά μα την κάναμε, το καθήκον μα το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει το καθήκον του. Και δεν θέλουμε να πάμε στο μπλοκάρισμα για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, να ενισχύσουμε τους πόρους μας χάρη σε αυτή τη δίκαιη φορολόγηση και να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη που θα χρειαστεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Κορμό ε, και κάποια άλλοι από την τον της λόγο. κύριο Λαγούτιου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχω όμως και τα τέσσερα λεπτά της Μαργαρίτας. Βλέπω ότι υπάρχει ενότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ 100% με τους πέντε πρώτους ομιλητές και χαίρομαι που είμαστε ενωμένοι στην επιθυμία μας να προχωρήσουμε. Έχουμε τρία προβλήματα εδώ. Την κύρωση από τα 27 μέρη, κράτη-μέλη του έκτακτου σχεδίου ανάκαμψη. Δεύτερον, να αποφύγουμε ε, νέα ύφεση όταν μετά από τρία χρόνια θα επανέλθουμε στο κανονικό προπολογισμό. Και τρίτο θέμα, να χρηματοδοτήσουμε την πράσινη συμφωνία. Αυτό το καλοκαίρι ήταν καταστροφικό για το κλίμα. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τη κύρωση, σε όλε τι χώρε λένε προσοχή, το Βέλγιο θα χάσει 12 δισεκατομμύρια, η Γαλλία θα χάσει 27 δισεκατομμύρια. Αν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ίδιους πόρους και ε, το Βέλγιο θα ανακτήσει 5 δισεκατομμύρια δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει τίποτα. 40 δισεκατομμύρια θα κερδίσει η Γαλλία και τίποτα δεν θα πρέπει ε, να επιστρέψει με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα για τους ίδιους πόρους. Νομίζω ότι έτσι η διεκδίκησή μας θα περάσει πιο εύκολα. Επίσης να αποτρέψουμε νέα ύφεση. Είμαι οικονομολόγο και παρακολουθώ εδώ και 30 χρόνια την Ιαπωνία. Κάθε φορά που σταματάει ένα μέσο ανάκαμψη, ξαναπέφτει στην ύφεση. Εδώ θα έχουμε μια, ε, ένα τριετή μηχανισμό ανάκαμψη. Αν όμω μετά τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να ε, επιστρέψουν στην λιτότητα, κινδυνεύουμε να υποπέσουμε σε μια ακόμη μεγαλύτερη ύφαση. Θα πρέπει λοιπόν μετά την τριετία να έχουμε σημαντικού πόρου, ιδιαίτερα το 2024 να έχουμε ένα πραγματικό κοινοτικό προπολογισμό που θα χρηματοδοτείται από ιδίου πόρου. Και τρίτον, για την πράσινη συμφωνία. Μια πραγματική πράσινη συμφωνία θα δημιουργήσει 5 εκατομμύρια θέσει απασχόληση παντού στον κατασκευαστικό τομέα, στη γεωργία, στην έρευνα, στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αν δεν έχουμε όμω μαζικέ και βιώσιμε κοινοτικέ επενδύσει, δεν θα δημιουργήσουμε ε, μια καλή δυναμική. Και χρειαζόμαστε ιδίου πόρου και μετά τα τρία έτη. Είναι σημαντικό το θέμα των ιδίων πόρων που θα το αποφασίσουμε σήμερα. Μία φορά κάθε 7 χρόνια ε, έχουμε λόγο στις διαπραγματεύσεις. Καλός ο Μόντι, αλλά τελικά ε, μας την έφεραν. Ε, θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους, στους διαπραγματευτές μας, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα συνδικάτα και να διεκδικήσουμε ιδίους πόρους. Επίσης, συμφωνία θέλουμε για το σύνολο του χρονοδιαγράμματος. Όλοι οι ίδιοι πόροι είναι σημαντικοί. Επίσης, μην ξεχνούμε το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που πρότεινε το 2011 ο Μπαρόζο. Και κάναμε υπολογισμούς και μπορούμε 50 δισεκατομμύρια το χρόνο να έχουμε παρά το Brexit και παρά την ε, οικονομική κρίση. Αν έχουμε δηλαδή κάθε χρόνο 50 δισεκατομμύρια ας πούμε 15 δισεκατομμύρια για να αποπληρώνουμε ε, τα 390 δισεκατομμύρια της επιχορηγήσης, θα μας μείνουν και πολλά χρήματα για το αέρασμο στην Πράσινη Συμφωνία και μόνο από το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα απεμπλέξουμε πολλά πράγματα. Για το φόρο για τα πλαστικά μπορούμε να πούμε ότι θα ξαναπέσει στους ώμους των πολιτών, για τον άνθρακα το ίδιο, αλλά ε, για το φόρο των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών ε, δεν θα πλήξει κάτι τέτοιο τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε ένα μικρό φόρο στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Την περασμένη εβδομάδα η Άγγελα Μέρκελ είπε ότι θέλει φέτος να καταλήξουμε στη συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε ζητώντας ένα τέτοιο συνολικό χρονοδιάγραμμα να είμαστε ισχυροί στη διαπραγματεύση και να ζητήσουμε και τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο κύριος και έχει το λόγο από το ECR. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Εδώ έχουμε φυσικά μία ε, καθυστέρηση. Ε, φαίνεται αυτό και στο μέσο ανάκαμψης και το ένα θεσμικό όργανο κατηγορεί το άλλο για αυτέ τι κολλησιεργίε, ε, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το καθεξής. Βέβαια, ε, θα έχουμε και τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα πρέπει να κυρώσουν την όλη διαδικασία. Ε, πολύ πρόσφατα είχαμε τα στοιχεία της Ευρωστάτ, της Ευρωστάτ και βλέπουμε ότι σε μερικές χώρες είχαμε μείωση του ΑΕΠ και κατά 20%. Και σε πολλές χώρες είναι πάνω από 10% η μείωση του ΑΕΠ, κάτι που προαναγγείλει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και ακόμη πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές οι μειώσεις γίνονται παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν δώσει δημόσιες ενισχύσεις ύψους 3-3 εκατομμύριων ευρώ, πολύ περισσότερα δηλαδή κονδύλια από τον επταετή προϋπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το μέσο ανάκαμψης και πολύ σύντομα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή η διελκυστίδα μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οι αλληλοκατηγορίες. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της παράτασης ε, του μέσου ανάκαμψης. Ένα τμήμα των επιχορηγήσεων ουσιαστικά θα μειώσει τα κονδύλια δύο βασικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Και αυτές οι δύο πολιτικές, κυρίως η, πολιτική, η αγροτική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική, μας εξασφάλισε την επιβίωσή μας στη διάρκεια της κρίσης και η, Γερμανία δικαίως ενίσχυσε τη γεωργική της πολιτική είναι δυνατόν, αναγνωρίζοντα τη σημασία μια τέτοια πολιτική και κατά τη διάρκεια τη πανδημία, να περικόπτουμε τόσο δραστικά τα κονδύλια τη κοινή γεωρική πολιτική. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κόκαλης από την ΚΟΕ, αυτή τη φορά προσωπώντα τον εαυτό του. Please, Mr. Kokali, can, you can uh, press your button. Αν θέλετε, κύριε Κοκάλη, να πατήσετε το κουμπί Speak. Ας περάσουμε στον επόμενο μιλητή και ίσως μπορέσουμε μετά να συνδεθούμε με τον κύριο Κόκαλη, ο κύριος Κίρτσος από το ΕΛΚ. We cannot hear you, Mr. Kirtsos. You have to... Δυστυχώς, κύριε Κίρτσο, δεν σας ακούμε. Θα πρέπει να πατήσετε το speak. Can you hear me? Με ακούτε? Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη πλειοψηφία ευρωβουλευτών επιθυμούν και προσπαθούν για ένα φιλοδοξότερο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι το Ταμείο Ανασυγκρότησης δεν είναι αρκετό για να ε, χρηματοδοτηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, όπως είπε ο συνάδελφος. Τα πράγματα πάνε χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Η εξακολούθηση της πανδημίας δεν μας επιτρέπει να οργανώσουμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το οριστικό τομέα ή ο τομέα των υπηρεσιών είναι πρωταρχική σημασία για την οικονομία. Κατά δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ένα δεύτερο κύμα COVID-19 και είναι προφανές ότι η πανδημία θα κρατήσει περισσότερο. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την ε, περίσταση αυτή. Και τρίτον, Διαρκώ καθυστερούμε σε σχέση με του ανταγωνιστέ μα, ε, την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Η Κίνα είναι πολύ αποτελεσματικότερη στην καταπολέμηση του COVID-19 και η ανάκαμψη τη κινέζικης οικονομία έχει διαρχίσει και οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική έχουν ε, πολλά προβλήματα μεν, αλλά είναι πολύ δυναμική ω προς την οικονομική του πολιτική και την αντιμετώπιση του COVID-19. Οπότε και θα πρέπει και εμεί νομίζω να προσπαθήσουμε να ακολουθούμε στον δρόμο των προτεραιοτήτων των περισσότερων των Ευρωβουλευτών, τη πλειοψηφία μας. Ευχαριστώ. Εδώ εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ε, αγορητών. Νομίζω θα ήταν λίγο να πούμε ότι το θέμα θα το ξαναδούμε σίγουρα, τουλάχιστον η διαπραγματευτική ομάδα, αλλά σίγουρα και η υπόλοιπη επιτροπή ε, στο σημερινό τη σχηματισμό. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το δούμε και στις επόμενες εβδομάδες σίγουρα, αναμφίβολα να σας θυμίσω εδώ την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με τον ε, Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μάλλον, τον κύριο Μάικλ Ροτ. Μίχαλ Ροτ. Να πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την πολιτική κτηρίων. Κάθε χρόνο τα θεσμικά όργανα πρέπει να αποβάλουν έκθεση για την κτηριακή τους πολιτική υπόψη της δημοσιονομικής αρχής. Στην Επιτροπή αυτή ήδη είχαμε συζητήσει με τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Βίλαντ και τον κύριο Σίλβα Περέιρα και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, για την κτηριακή πολιτική του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την προσέγγιση για την κτηριακή πολιτική και τα βασικά έργα που έχουμε μπροστά μας. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μαρκ Μπεκέτ, διευθυντή του Γραφείου Υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Τόμας Κίρχνερ, ο οποίος είναι υπεύθυνο της Υπηρεσίας Υποδομών και Κτηρίων του Λουξεμβούργου. Έχετε το λόγο κύριε Μπακέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ίσως δύο λόγια για το συνολικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα προ... Ε, χαρτοφυλάκιο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ε, από τα οποία ένα σύνολο μάλλον ε, ενό εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, των οποίων 907.000 είναι γραφεία και 50 περίπου κτίρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 60% είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 40% είναι από αυτά που μισθώνονται, όπω για παράδειγμα στην Όλαφ. Ε, το πλαίσιο για την ε, κτηριακή μας πολιτική ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε κάποιες περιπτώσεις παράτασης ή επαναδιαπραγμάτευσης κάποιων επιμισθωμάτων, συμβάσεων και θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες επιφάνειες και εκτάσεις σε ιδιωτικά κτίρια για να είναι πιο αποτελεσματικά και από την άποψη της ενέργειας. Και βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις επιφάνειες που ήδη διαθέτουμε. Η προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει για το Κοινοβούλιο ε, για το θέμα ε, αυτό ήταν ε, πέρυσι στις 24 Σεπτεμβρίου και έκτοτε φυσικά το όλο σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά. Έχουμε ένα σκηνικό σχεδόν κατόπιν της πανδημίας από το οποίο έχουμε αντλήσει μια σειρά από διδάγματα και έχουμε και τις φιλοδοξίες του Green Deal που θα πρέπει να ε, όπως προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Τροπή, θα πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε ουδέτεροι προς τη χρυσή άνθρακα μέχρι το 2030 και βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του πολιτικού του μουσιονομικού πλαισίου. Οι άξονε για δράση μα είναι να χρησιμοποιήσουμε με περισσότερο τρόπο κάθε τετραγωνικό μέτρο και με τρόπο πιο ευφύω προ την ενέργεια. Τώρα, ε, κάναμε μια ε, ταχεία ανάλυση του ποιε είναι οι απειλέ αδυναμίε, ευκαιρίε και τα δυνατά μας σημεία σε σχέση με τα θέματα αυτά. Τα βλέπετε στη διαφάνεια, δεν θα περάσω τις λεπτομέρειε, για να ε, μην εξαντλήσω το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Τα έργα που θα, σας υποβληθούν στην κρίση σας στο μέλλον. Από τη μια, η ανακαίνιση του Αλμπέρ Μπορσέτ, του Κέντρου συνεδρίου Ραλμπερ Μποσέτ. Μιλάμε εδώ για, επίσης για ανακαίνιση του ΛΟΑ 51, ένα πρόγραμμα μίσθωσης για τον Πολιό 159. Ε, αυτά είναι σε ματοπατική φάση για ταυτόχρονα και ε, διεύρυνση του κτηρίου Μοντουαγέ 34. Ένα κτίριο που θα το αφήσουμε για να πάμε σε καινούργιες εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά τα οποία σκεφτόμαστε, κυρίως την, ε, τον σταθμό Palmerston, επίσης μια νέα ανάπτυξη των κτηρίων Μπρεντέλ και Μπρεντέλ 2 και μετά μια νέα ανάπτυξη των κτηρίων της περιοχής Μπολιέ, των Μπολιέ 23, 31 και 33. Ταυτόχρονα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με το κτίριο Λουά 130, αλλά αυτό έχει ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εκεί θα πρέπει να δούμε και κατά πόσον θα υπάρξει και μια νέα κανονικότητα ε, και πώς θα διαμορφωθεί αυτή μετά την κρίση του COVID. Τώρα για τα έργα που ήδη σας ανέφερα, τα βλέπετε στην διαφάνεια, το ίδιο και για τα μελλοντικά σχέδια. Μερικά στοιχεία για το πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα τετραγωνικά που διαθέτουμε με τρόπο πρασινότερο και ευφιέστερο. Όπως βλέπετε, κάθε τετραγωνικό ε, κτηρίων υψηλών επιδόσεων θα μας επιτρέψει να έχουμε μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά ταυτόχρονα να περιορίσουμε και το σύνολο των επιφανειών που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε κάποιες χιλιάδες ε, λιγότερο, ε, περισσότερο μάλλον σε πάρκα τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα πραγματικότητα και πώς θα υλοποιήσουμε και νέες μεθοδολογίες που έχουμε στην διάθεσή μας. Η τελεεργασία θα λάβει σημαντικότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν και αυτό θα επηρεάσει και τη χρήση των επιφανειών που διαθέτουμε. Να αναφέρω εδώ δύο στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την νομοθεσία που ισχύουν στην πόλη των Βρυξελών. Πρώτα απ' όλα ο νόμος ΠΛΑΣ που έχει να κάνει με τη μείωση των βασικών εκπομπών σε σχέση με την κατανάλωση ε, ενέργειας από τα κτίρια. 10% προβλέπεται μείωση στο 2025. Αυτό επηρεάζει ότι θα κάναμε κάποια από τα κτίρια μας που είναι πολύ παλιά για να περάσουμε σε κτίρια καινούργια με καλύτερες επιδόσεις και μετά ο νόμος Κομπράς για τη μείωση των ε, ε, χώρων σταθμ, των χώρων στάθμευσης. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μετατροπή κάποιων ε, γκαράζ, κάποιων χώρων στάθμευσης, με την φιλοδοξία να δημιουργήσουμε ένα hub, ένα κέντρο παρκαρίσματος για ποδήλατα. Ε, λόγω του περιορισμού στον χρόνο τη ομιλία μου, θα ήθελα να σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε και με στη διάθεσή σα για περαιτέρω ερωτήσεις και απαντήσει. Ευχαριστούμε κύριε Μπεκέτ, ο κύριο Κίσνερ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας παρουσιάσω την ε, κατάσταση για το Λουξεμβούργο. Έτσι όπως αναφέρθηκε η σχέση με τις ε, Βρυξέλλες, ε, πολλά έχουν συμβεί από τον περσινό Σεπτέμβριο, πράγμα το οποίο θα έχει και επιπτώσεις για τα όσα θα συμβούν στο μέλλον και στο Λουξεμβούργο. Σε ό,τι αφορά τα ίδια τα κτίρια δεν θα είναι τόσο μεγάλε οι επιπτώσεις. Αντιθέτως, οι επιπτώσει θα αφορούν στη χρήση και τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κτίρια. Καταρχήν, να σα υπενθυμίσω εν συντομία πώ έχουν τα πράγματα τη σήμερα ημέρα στο Λουξεμβούργο σε ό,τι αφορά τα κτίρια. Έχουμε λοιπόν 4.700 ε, άτομα ως ε, προσωπικό, ε, κατανεμιμό σε 17 κτίρια γραφείων ε, σε τρία διαφορετικά σημεία της ε, πόλης, ε, Κάσπερ, Κίσπερ και κέντρο της πόλης. Όμως επειδή μέσω πρόθεσμα θα περάσουμε σε ένα νέο κτίριο στο Ζαμονέδιο, τα περισσότερα από τα κτίρια μας είναι μισθωμένα, εκτός από το Euroforum, το οποίο έχει τεθεί σε μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική δηλαδή μίσθωση. Όπως γνωρίζετε, το Ζαν ε, Μονέ αποτελεί την απαρχή, αν θέλετε, το βασικό πρόγραμμα για μας στο Λουξεμβούργο. Ε, βρίσκεται ακριβώ στο, στο Κίρχπερκ, σε αυτή την ε, γειτονιά και ο συνολικός προπολογισμό είναι 442,8 εκατομμύρια ευρώ με 3.700 θέσει εργασία. βασικά πολύ σημαντικό ε, εδώ είναι το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας ε, του κτηρίου. Ε, θα λάβει λοιπόν την αξιολόγηση BRIM ως εξαιρετικές επιδόσεις σε αυτό το τομέα. τώρα, οι εξκαφικές εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τον Ιούλιο. Θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες στις επόμενε διαφάνειες οι φάσεις τώρα 1 και 2 σε ό,τι αφορά δηλαδή, την κατασκευή έχουν ξεκινήσει και να σας πω σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα ότι ε, για τη φάση 1 η οποία αφορά στο σε κτίριο, το οποίο βλέπετε εδώ και στη φωτογραφία, αρχικά λοιπόν έχει προβλεφθεί η ε, παράδοση ε, για τον Φεβρουάριο του 2023 και από εκεί για τη δεύτερη φάση μέσα στο 2024. Βέβαια τώρα με το COVID αλλά και επειδή υπήρξαν και κάποια άλλα ζητήματα είχαμε για κάποιες ε, περιπλοκές καταρχήν έκλεισε ε, για ε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντελώ το εργοτάξιο και μέχρι και σήμερα η παραγωγικότητα στο εργοτάξιο έχει μειωθεί γιατί χρειάστηκε να εφαρμοστεί ένας νόμος τρόπος εργασίας και να ληφθούν νέα προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό. Και βέβαια όλα αυτά έχουν επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα ε, ολοκλήρωση, αλλά και στον ε, προπολογισμό που θα χρειαστεί εν λόγω επιπτώσει να, να αξιολογηθούν. Δεν ε, μπορώ όμω να σα δώσω περαιτέρω λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ ε, πρόωρα τα πράγματα. Δεν έχει δηλαδή ακόμα περάσει βέβαια και η κατάσταση και δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα όλε τι πληροφορίε. Η ε, Επιτροπή Καθοδήγηση στο Steering Committee ε, θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα αυτή η GMO Steering Committee η οποία συνέρχεται και με τους διαχειριστές του προγράμματος δηλαδή τις αρχές του Λουξεμβούργου εδώ προκειμένου ακριβώς να συζητηθεί το ζήτημα αυτό μεταξύ άλλων δηλαδή ο αντίκτυπος από το COVID-19 αλλά θα συζητηθούν και άλλα τεχνικά θέματα τα οποία έχουν τεθεί από την πλευρά του αρχιτέκτονα. Όταν λοιπόν τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα ω προ τι επιπτώσει του COVID σε επίπεδο προπολογισμού και χρονοδιαγραμμάτων, θα σα ενημερώσουμε. Τώρα, Όπω σα είπα, ότι θα έδειξα κάποιε φωτογραφίε. Τον ε, Ιούλιο του 2019 βλέπετε εδώ μια φωτογραφία, ε, πριν ένα χρόνο δηλαδή, που έχουν ξεκινήσει εξαφικέ εργασίε. Και βλέπετε εδώ ε, στην κάτω πλευρά και κάποια ε, ακόμα κατάλοιπα από το προηγούμενο ε, Ζαμονέ. Και τώρα μια νέα φωτογραφία από τον Ιούνιο του 2020 όπου έχουν προχωρήσει εργασίες. Και ειδικότερα στο κάτω κομμάτι βλέπετε ε, το πώς προχωράει η φάση 1 σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εργασίες κατασκευής περισσότερο. από εκεί και μετά να σας πω ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε μία σειρά από τις συμφωνίες εμεί στο που έχουμε σε ό,τι αφορά το Ζαμονέ, γιατί για κάποιες από αυτές ε, ήδη έχουμε ε, λάβει την έγκριση από την ε, αρχή προπολογισμού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κτίρια Μπέχε και Αριάν σε ό,τι αφορά δηλαδή και τι ε, ε, ημερομηνίε μετακόμιση, αλλά και σε ό,τι αφορά την απαραίτητη ευελιξία που θα πρέπει να προβλέψουμε σε ό,τι αφορά ακριβώ την περίοδο αυτή τη μετάβαση. Από εκεί και μετά ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα τη λειτουργία του διοργανικού κέντρου, δηλαδή βερφονιπιακού σταθμού, το International Children's Center, το οποίο τη σήμερα ημέρα θεωρείται ως αρκετά σε εκτίριο. Θα υπάρξει μια πρώτη συζήτηση σε επίπεδο της αρχής προπολογισμού ε, στα τέλη αυτού του έτους ε, και από εκεί και μετά ένα ακόμα ζήτημα είναι το ταχυδρομικό κτίριο του Μέρσια, το οποίο θα λάβει μια επιστοποίηση από έναν ε, φορέα, των DGMB, ο οποίος πραγματικά θεωρείται ότι δίνει εξαιρετικές επιστοποίησεις και εκείνος από την πλευρά του και όλα αυτά λοιπόν είναι τα όσα αναμένουν. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ, μόνιμη συγκεντρία για τα θέματα της κτηριακής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Μπεκέτ ε, από το γραφείο των Βρυξελών, τον κύριο Κεσνέρα από το γραφείο των Βρυξελών, του Λουξεμβούργου, συγγνώμη, που παρακολουθούν το θέμα τη κτηριακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό. Μερικέ ερωτήσει, οι οποίε έχουν σχέση και με όσα μα παρουσιάσατε, αλλά και για να σα ζητήσω κάποιε διευκρινήσει. Αναφέρατε τους στόχους του Green Deal, τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για τα έργα της εργασίας που πρόκειται να ξεκινήσουν για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Ιδίως για αυτούς που πολιτικώς έχουν τεθεί από τα θεσμικά μας όργανα ή και από τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Ε, όλος ε, για τις Βρυξέλλες διαπιστώνω, όπως και πολλοί συνάδελφοι, ότι πολύ συχνά ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι πρώτα απ' όλα να γκρεμίζουμε κτίρια, ακόμα και κτίρια που είναι μόλις 30 ετών. Ε, κάτι που έχει συμβεί για το ΛΟΑ 130, ένα μεγάλο εργοτάξιο της Επιτροπής της Βρυξέλλης. Έχετε τρόπο να χρησιμοποιείτε λίγο λιγότερο αυτό το σύστημα ε, των ε, κτηρίων που είναι έτσι σύντομης διάρκειας ζωής δεν είναι πολύ βιώσιμο αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα που με ενδιαφέρει, δεν μας είπατε πολλά γι' αυτό, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Ε, η πανδημία του COVID μας ε, ανάγκασε να εργαζόμαστε διαφορετικά. Είναι πολλοί πλέον όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως. Νέοι τρόποι διοργάνωσης της εργασίας ε, αρχίζουν να επιβάλλονται το open space και η οργάνωση τη εργασία γενικώ είναι θέματα που θα μα απασχολήσουν ε, και το τι μορφή θα πάρουν στο μέλλον. Είπατε για μείωση 25% της επιφάνειας ε, στις Βρυξέλλες. Ε, έχετε κάτι υπόψη πιο συγκεκριμένο, πιο διοργανωμένο πώς θα επηρεάσει αυτή η κρίση τον τρόπο που εργαζόμαστε και τέλος και τα κτίρια που χρησιμοποιούμε. Και δύο πολύ πρακτικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά το έργο ΛΟΑ 130, ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο βεβαίως θα ξεκινήσει το 2025, αλλά για το οποίο ο διαγωνισμός μεταξύ αρχιτεκτόνων σχεδιαστών έγινε ήδη πέρσι. Πότε προβλέπετε να υποβάλλετε στην Επιτροπή μας αυτό που ονομάζουμε την έγκαιρη ειδοποίηση, το early warning, για να εξετάσουμε το έργο αυτό και να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε και το κατά πόσον είναι ορθό το κόστος του. Και μετά για το Λουξεμβούργο και το έργο Ζαμονέ θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα, να μας ε, πείτε πόσο θα κοστίσει η καθυστέρηση του έργου. Ένα έργο ε, επίσης πολύ μεγάλο, 440 ε, εκατομμύρια ε, είναι όσο θα κοστίσει. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλερ και τώρα σκιώδεις εισηγητές. Για δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Χολμάγερ δεν είναι εδώ, οπότε ο κύριος Ούζακοφς, ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν αναφερόμαστε σε ζητήματα κτηριακής ε, ε, πολιτικής, ε, έχουμε, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον κανένας μας εδώ στην Επιτροπή των Προπολογισμών, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στο μέλλον κάτι κάθε φορά που υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα του προπολογισμού ενό ε, έργου, να λαμβάνουμε ε, πληροφορίε εγκαίρω, ε, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Κούστορα, ID. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα από την πλευρά μου. Αναφέρθηκε ε, ότι οι επιφάνειες θα μειωθούν από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα σε 743.000 743 ε, τετραγωνικά μέσα. Οπότε εγώ σας ερωτώ πώς θα το επιτύχετε αυτό συγκεκριμένα θα εφαρμόσετε δηλαδή ε, όλες αυτές τις νέες δυνατότητες τηλεργασίας ή θα υπάρξουν και άλλες προσαρμογές και σε ποιο βαθμό έχετε προχωρήσει σε ό,τι αφορά αυτή τη μείωση. Μετά, ε, κάτι άλλο, αναφερθήκατε στο ότι θα πρέπει να μειωθούν ε, οι δαπάνε κατανάλωση λειτουργία δηλαδή των κτηρίων κατά 10%. Οπότε και σε σχέση με αυτό σα ερωτώ πώ θα το επιτύχετε συγκεκριμένα. Ε, και επίσης δεν είναι πολύ βραχυπρόθεσμος αυτός ο ε, στόχος, ε, δηλαδή εάν πραγματικά έχουμε μια ανακατασκευή τέτοιων κτηρίων όπως τον Τζαν Μονέ, τότε δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό να επιτύχουμε υψηλότερη μείωση, δηλαδή όχι μόνο 10%. Και από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τα Joint Research Centers, κοινά λοιπόν, αναφέρεται εδώ ότι ε, πρόκειται για ένα, ε, μια υπηρεσία ακριβώς ε, ε, επιστημονική και ερευνητική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ο στόχος είναι να συμβάλλει στους γενικούς στόχους του Horizon 2020. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμμετέχει, αν θέλετε, από τη δική της πλευρά στο, στο Horizon. 10 ε, δισεκατομμύρια στο πλαίσιο του Horizon ε, διανέμονται στα διαφορετικά κράτη-μέλη, ε, προκειμένου ακριβώ να γίνουν επενδύσει στον τομέα τη επιστήμη και προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία. Εάν όμω τελικά έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή εάν έχουμε να κάνουμε με κτίρια τη Επιτροπή διατίθενται για την επίτευξη και την πρόθεση των στόχων του Horizon, τότε δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Δεν υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή δεν γίνεται η χρηματοδότηση εδώ λανθασμένων στοιχείων, δηλαδή με κονδύλια του Horizon χρηματοδοτείται τελικά η λειτουργία κτηρίων της ίδιας της Επιτροπής. Ε, κάτι ίσως να μην κατάλαβα εδώ σωστά. Ευχαριστούμε. Ε, κύριος Αντρέσεν τώρα ε, για τους πράσινους. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά ε, την στρατηγική, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το να επιτύχουμε ουδετερότητα, σε ό,τι αφορά το, ε, τη χρήση του άνθρακα, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ένας άλλος συνάδελφος, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενημέρωση, ότι καλό θα είναι και απαραίτητο να λαμβάνουμε εγκαίρως την πληροφόρηση σε ό,τι αφορά ε, τα νέα project και το τι συμβαίνει και τις αλλαγές σε σχέση με αυτά. Γιατί εδώ μέσα σε αυτόν τον πρώτο χρόνο που συμμετέχω στις εργασίες του Κοινοβουλίου έχω διαπιστώσει ότι συχνά δεν έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια ζητήματα γιατί ακριβώς τα ε, project θεωρούνται επίγοντα και έκτακτα αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τη φύση των αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά εδώ αυτό το τομέα της εκτηριακής πολιτικής. επάνω σε ό,τι αφορά τη στατική για την ουδετερότητα άνθρακα, να πω ότι αναφερθήκατε σε κάποιες ε, ε, αλλαγές συμπεριφορικές, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τον τρόπο εργασία. Οπότε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ε, τι ακριβώς εννοείται εδώ, δηλαδή πέρα από τα bicycle hubs, αυτά τα κέντρα λέγεις για, για τα ε, ποδήλατα, θέλετε να κάνετε και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το ενεργειακό ζήτημα, γιατί νομίζω πως τα όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωση έχουμε και ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά και τα απόβλητα, οπότε θέλετε να κάνετε και σε σχέση με τα απόβλητα και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ε, κατανάλωση ενέργεια, θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς θα κάνετε για να επιτευχθεί αυτή η ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τον άνθρακα ως το 2030. Υπάρχουν δηλαδή μια, φορά από μια σειρά από διαφορετικά στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας, οπότε θα ήθελα να μου πείτε με λίγη παραπάνω λεπτομέρεια τι ακριβώ. Σας ευχαριστώ. κύριο Ζόνιτσα, εκ μέρους του ECR. Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε την κυρία Κέλλερ, την εισηγητριά μας. Ε, είδαμε ε, τα, κτίρια και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία. Τι γίνεται με αυτές τις κίτρινους σωλήνες που φέρουν φυσικό αέριο στα κτίρια. Υπάρχουν τέτοια σχέδια, πόσο θα κοστίσουν. Επίσης, ε, γίναμε μάρτυρες μιας μετάβασης ε, στην τηλεργασία. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες ο καθένας, αλλά μήπως ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε τώρα αν ε, έχει νόημα ε, αντί να ε, επενδύουμε σε κτίρια που τα εγκαταλείπουμε λόγω της πανδημίας, να αφιερώσουμε ε, κάποιους δημοσιονομικούς πόρους για την τελειοποίηση του συστήματος της τηλεεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζόντσα. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο από την Ομιγύρη ή από τους εξαποστάσεως συμμετέχοντες. Οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στους καλεσμένους μας, τον κύριο Μπεκέ και τον κύριο Γκίρχερ, για να απαντήσουν στις πολυάριθμες ερωτήσεις που τέθηκαν. Ο κύριος Μπεκέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω τις ερωτήσεις για να κερδίσουμε και χρόνο. Σε ό,τι αφορά τη νέα πράσινη συμφωνία, όπως είπα, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε τις εκπομπές μας και φυσικά θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε και την ε, ενεργειακή μας κατανάλωση. Γιατί η πιο φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνουμε. Επίσης, θα, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ε, στα θέματα της κινητικότητας, για να έχουμε μια πιο ήπια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα απόβλητα. Και εκεί θα έχουμε σημαντική ενίσχυση για να περιορίσουμε τα απορρίμματα, να έχουμε μια καλύτερη διαλογή και κατάλληλους κλάδους ανακύκλωσης. Γιατί σε λίγες μέρες με την κρίση της πανδημίας COVID ε, εγκαταλείψαμε το χαρτί. Γίναμε όλοι πέπερλες. Γιατί να επανέλθουμε σε μαζική χρήση χαρτιού, αφού συνηθίσαμε να μην το χρησιμοποιούμε. Επίσης, ε, ε, σε ό,τι αφορά και την καντίνα, το self-service, ε, τις καφετερίες και εκεί προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Σε ό,τι αφορά την ε, έγκαιρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ε, επισήμανα τα θέματα που θα σας υποβάλλουμε τους επόμενους μήνες, ώστε να μην υπάρχει κανένας ευνηδιασμός ή καμία έκπληξη που ανέφεραν κάποια μέλη της Επιτροπής, Ήδη τα προαναγγείλαμε. Σε ό,τι αφορά τις νέες μεθόδους εργασίας, ε, γίνεται αυτή τη στιγμή κάποια αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης COVID και στην τηλεργασία και στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας που επιτρέπουν μια αποτελεσματική τηλεργασία, όπως φάνηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, σκεφτήκαμε πώς να εξοπλίσουμε τους συναδέλφους ώστε να μπορούν να τηλεργάζονται από την οικία τους με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχίζεται η σχετική συζήτηση. Επίσης, πιο ορθολογική χρήση των κτηρίων με λιγότερα τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιούμε. Και εκεί θα κάνουμε κάποια οικονομία και ένα τμήμα των οικονομιών που θα κάνουμε από την μικρότερη χρήση των τετραγωνικών μέτρων θα τα θα χρησιμοποιήσουμε για να εξοπλίσουμε καλύτερα τους συναδέλφους για να τηλεργάζονται. Θα πρέπει όμως να αφήσουμε, ε, να αφήσουμε άθικτο τον κοινωνικ, τους κοινωνικούς δεσμούς, να αποφύγουμε την απομόνωση. Και εκεί θα πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία. Αλλά όλα αυτά τα εξετάζουμε. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους ε, κατασκευής, Όντως, για μερικά κτίρια έχουμε συνηθίσει να έχουμε μία ωφέλιμη διάρκεια χρήσης 30 ετών. Και οι εργολάβοι είτε ε, κρατούν απλώς το σκελετό του, το, του κτηρίου, τα θεμέλια, τις στήλες και μετά το επανεδύουν, επανεξοπλίζουν ώστε να γίνει καλύτερο από ενεργειακή άποψη. Αλλά πολύ συχνά δυστυχώ προβαίνουμε σε πλήρη κατεδάφιση του κτηρίου. Όλα τα θεσμικά όργανα το κάνουν, αλλά για εύλογου λόγου, πολλές φορές. Θα σας δώσω το παράδειγμα του πύργου, ε, πύργου 1 που ε, βρίσκεται στη θέση ενός παλιού ξενοδοχείου. Δεν μπορεί το ξενοδοχείο να το μετατρέψουμε σε κτίριο με γραφεία λόγω του, του ύψους που έχουν οι οροφές. Οπότε στις Βρυξέλλες ε, τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι προσάρμοστα, να μην είναι μόνο γραφεία ή μόνο κατοικίες ή μόνο καταστήματα. Να μπορούν να περνούν από τον ένα τρόπο χρήση στον άλλο. Αυτό προβλέπει η νέα ε, στρατηγική για τις Βρυξέλλες. Επίσης για το κτίριο ΛΟΑ 130. Όταν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το μέλλον του σχεδίου ΛΟΑ 130, θα έρθουμε εγκαίρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας ενημερώσουμε για τις προθέσεις μας ως προς το σχέδιο για το ΛΟΑ 130. Προς το παρόν είναι πρόωρο κάτι τέτοιο, γιατί συνεχίζονται ακόμη οι συζητήσεις και οι μελέτες. Δεν έχουμε καμία ακόμη προπτική ιδέα για το τι θα γίνει με το ΛΟΑ 130, για να σας ενημερώσουμε. Σε ό,τι αφορά τα κτίρια του Κοινού Κέντρου Ερευνών, ένα μικρό του προσωπικού, 200 περίπου υπάλληλοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες για μια γενική διεύθυνση που έχει πάνω από 2.000 απασχολούμενους εργαζόμενους. Έχουμε μια δραστηριότητα που αφορά τον ορίζοντα 2020, αλλά δεν χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του ερευνητικού προγράμματο. Πρόκειται για κτίρια που χρηματοδοτούμε εμεί από την μελλοντική στήλη 7. Δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Απλώ προσφέρουμε γραφεία στους ερευνητέ του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Α, για, τα, για το 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα ε, αυτή είναι η συνολική επιφάνεια, το συνολικό εμβαδόν, το 1 εκατομμύριο μέτρα, αλλά έχουμε πολύ λιγότερα τετραγωνικά μέτρα ε, για τα γραφεία και ιδιαίτερα ε, τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. έχουμε 795.000 τετραγωνικά μέτρα. Ε, θα τα μειώσουμε κατά 50.000 τετραγωνικά μέτρα μέχρι το 2024. Οπότε, θα περιοριστούμε σε 745.000 τετραγωνικά μέτρα. Αν με του νέου τρόπου εργασία και από τα διδάγματα που θα αντιλήσουμε από την πανδημία COVID, αν αντιληφθούμε ότι μπορούμε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο ε, το εμβαδόν των γραφείων, θα το κάνουμε. Και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως αν γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι κάλυψα το σύνολο των ερωτήσεων και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Μπεκέρο. Ο κύριο Κίρχινερ έχει το λόγο. Ε, για να επανέλθω σε ερωτήσεις. Καταρχήν για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εγώ αναφέρθηκα στα δύο πιστοποιητικά, στον BREAB και στο DGMB. Πρόκειται για πιστοποιητικά που αφορούν την βιωσιμότητα των σχεδίων, τη διάρκεια και όλες τις φάσεις από τη σύλληψη, την κατασκευή μέχρι το τέλος ζωής ε, του κτίριου. Και υπάρχουν διάφορα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση. Αφορούν την ε, διαχείριση, την ενέργεια, τη μεταφορά, το, την υδροδότηση, τα υλικά, τα απόβλητα και η χρήση του εδάφους, αλλά και η οικολογία. Πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο που χαρακτηρίζει τις ε, ε, επιδόσεις των μελλοντικών κτίριων. Σε ό,τι αφορά την πανδημία COVID και τον αντίκτυπό της στον τρόπο εργασίας, δεν έχουμε ε, διαφορά ε, Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες. Έχουμε κοινή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διάφορα γραφεία και στις δύο έδρε. Προσπαθούμε να δούμε τις επιπτώσεις ε, που θα έχει ο νέος τρόπος εργασίας στη χρήση των κτηρίων μας. Από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί το κτίριο Ζαμονέ, θα μας μείνουν τρία ακόμη κτίρια για, με γραφεία, το Ζαμονέ 2, το Euroforum και το κτίριο για την υπηρεσία εκδόσεων. Και μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε πολύ λιγότερο χώρο για τους υπαλλήλους που θα στεγαστούν στο Ζαμονέ 2 γιατί πολύ περισσότεροι θα εργάζονται σε τηλεργασία. Και θα δούμε με τι μέτρα θα μπορέσουμε ε, να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το εμβαδόν ε, στο Euroforum ή στην υπηρεσία εκδόσεων. Κατά πάσα πιθανότητα στο Euroforum γιατί είναι και το παλιότερο κτίριο που έχουμε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον. Ήδη έχουμε αρχίσει την εξέταση και από τη στιγμή που θα διαμορφώσουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα για το νέο τρόπο εργασίας και το συγκεκριμένο ε, αντίκτυπο της πανδημίας στη χρήση των γραφείων θα επανέλθουμε. Σε ό,τι αφορά το κόστος της καθυστέρησης. Εγώ σας έδωσα τις τελευταίες ημερομηνίε και χρονοδιαγράμματα. Μάλλον θα υπάρξουν αλλαγές. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να ποσοτικοποιήσουμε αυτή την ολιγόρια. Γιατί ακόμη και μετά την καθυστέρηση έχουμε κάποια μέσα εκ των υστέρων για να υπολογίσουμε το οικονομικό κόστος. Ένα τμήμα του κόστους αφορά φυσικά την κατασκευή και ένα άλλο την στέγαση των υπαλλήλων για τους επιπλέον μήνες όσο καθυστερεί το έργο. Αυτά και νομίζω ότι ολοκλήρωσα τα στοιχεία για το Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Κυρία Κέλλερ. Θέλετε το λόγο για κάποια τελικά σχόλια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Μπεκέρ και κύριε Κύρχινερ για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους, τους και οδησηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που υπέβαλαν. Ε, λίγες συμπληρωματικές σκέψεις. Ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του, της πανδημίας COVID ε, στις, στους, στον τρόπο εργασίας, τηλεργασία και νέα οργάνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ε, ενημέρωσε ότι υπάρχει μια νέα διοργανική ομάδα σε μια παρόμοια ακρόση που είχαμε τον Ιούλιο. Εγώ θα σας πρότεινα να μας στέλνετε που και που ε, τις σκέψεις και την πορεία των εργασιών σας για το νέο τρόπο εργασίας σε μια λογική φυσικά που εξαρτάται από το κάθε θεσμικό όργανο, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά καλό είναι να έχουμε μια ανταλλαγή ε, πρακτικών ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Σε ό,τι αφορά το κτίριο ΛΟΑ 130, 100.000 τετραγωνικά μέτρα είναι το συγκρότημα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε από τώρα να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα, γιατί ε, νομίζω ότι η συγγραφή υποχρεώσεων έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έγινε το 2018. Και πριν από ένα χρόνο ανατέθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο ε, αρχιτεκτόνων μετά τη συγγραφή υποχρεώσεων. Μας λέτε ότι είναι πρόωρο, αλλά κάποιες αδρές γραμμές του σχεδίου θα πρέπει ήδη να τις έχετε και κάποια προοπτικές για το κόστος. Και γι' αυτό έχουμε την έγκαιρη προειδοποίηση, όχι αφού ε, οριστικοποιηθεί το σχέδιο. Έγκαιρη προειδοποίηση έχει νόημα σε μια προηγούμενη φάση, όταν ξεκινά το πρόγραμμα και όχι όταν ολοκληρώνεται το σχέδιο. Σε ό,τι αφορά επίσης τη μέθοδο κατασκευής που έχει σχέση με τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Εγώ θα ήθελα στην ανάλυση των φακέλων να περιλάβετε ε, και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για επαναχρησιμοποίηση των ε, υπαρχών των κτίριων. Γιατί και το θέμα των αποβλήτων είναι σημαντικό στο καλάθι των αποβλήτων, τα απόβλητα της, του κατασκευαστικού κλάδου είναι πάνω από τα, το 50% των συνολικών απορριμμάτων. Οπότε γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε, να μην ζητήσουμε επαναχρησιμοποίηση των κτίριων που ήδη, υπάρχουν. Γιατί δυστυχώς οι εργολάβοι προτιμούν να καταδαφίζουν και να ξαναρχίζουν από την αρχή. Με βάση μια νέα συγγραφή υποχρεώσεων και επίσης περιμένουμε την αξιολόγηση του συμπληρωματικού κόστους για το Ζαν Μονέ λόγω της καθυστέρησης και λόγω του επιπλέον κόστους που θα χρειαστεί για την παράταση κάποιων μισθωτηρίων συμβολέων για να παραμείνουν οι υπάλληλοι όσο δεν μπορούν να μετακομίσουν στο Ζαμονέ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη διαφάνεια και την ενημέρωση που μας κάνατε. So I Επαναλαμβάνω, μερσή, ευχαριστούμε ε, για όλους για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι ο χρόνος ε, για τις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της πρώτης ε, συνόδου, της χθεσινής, των χθεσινών ψηφοφοριών μεταφορά των ε, ε, ποσών Γενικός Προπολογισμός 2020. Ε, η κυρία Μόνικα Χολμάγερ επέφθηνε για την γνωμοδότηση ΔΕΚ 15-2020 εγκρίθηκε και επίσης μεταφορά των ταμιεύσεων Γενικός Προπολογισμός 2020 η κυρία Καρδία Σαμπάλ για τα υπόλοιπα τμήματα. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ε, ιδίες πρωτοβουλίας 1-2020 και ΔΕΚ 1-2020 εγκρίθηκε και ε, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο VAB 05T20 ε, και VAB 06α20 εγκρίθηκε για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωζέ Μανουέλ Φερνάντες και Βαλερή Αγέρ. Ε, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν είναι η ε, συμβαστική H, J, I, K η τροπολογία 21, η συμβιβαστική L, η τροπολογία 22, η τροπολογία 23, 24, η συμβιβαστική M, η συμβαστική Α, η συμβαστική B, η τροπολογία 3, η συμβαστική C, η συμβαστική D, η συμβαστική Ε, η συμβαστική F, η συμβαστική G, η συμβαστική GA, η 9, 10, 12, 13, συμβαστική GB. Τροπολογίες που απερίφθησαν 115, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 139, 140, 149, 152, 153, 30, 32, 31, 43, 45, 48, 65, 66, 67, 68, 74, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103. Τώρα, το πρόγραμμα Youth for Health του κυρίου Στεφανούτα. Τροπολογίε που εγκρίθησαν. Συμβαστική 1, συμβαστική 2, συμβαστική 3, τροπολογία 79, τροπολογίε που απερίφθησαν 95, 55, 57, 58, 68, 14. Πρόγραμμα Reactive, Κάρλο Ρέσλερ. Τροπολογίες που εγκρίθησαν το μπλοκ 1, ε, το μπλοκ 2 και το μπλοκ 3 η τροπολογία 56, συμβαστική 1, 2. Η τροπολογία 71, ε, η τροπολογία 88, 16, 96, 18, 17, 19, 1. Συμβαστική 3, 29, συμβαστική 4, 37, 38, 39, 40, συμβαστική 5, συμβαστική 6, συμβαστική 7, συμβαστική 8, τροπολογία 6. Τροπολογίες απερίφθησαν είναι η 76, 89, 92, 94, 27, 30, 31, 32, 43, 51. Ο Ενωσιακό ε, Μηχανισμό Πολιτική Προστασία του κ. Χέρμπ, τροπολογίε που εγκρίθησαν, ε, τροπολογία 45, συμβαστική 5, τροπολογία 49, 50, 54, 52, 4, 53, 55. Συμβαστική 6, τροπολογία 6, 7, 58, 8, 9, 10, 60, 12. Συμβαστική 1, τροπολογία 15, 12. Συμβαστική 1, τροπολογία 15, 17. Συμβαστική 2, τροπολογία 23, 24, 27. Συμβαστική 3, συμβαστική 4, τροπολογία 34, 36, 37, 1, 2, 39, 41, 43, 44, 3. Τροπολογίες απερίφθησαν. Τροπολογία 51, 56, 59, 18, 25, 26, 28, 35, 38, 40, 42. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για αυτήν την άκρος ενδιαφέρουσα και συναρπαστική στιγμή της συνεδρίασης. Ευχαριστώ, το εκτιμώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει τώρα να περάσουμε στις προφορίες και να ελέγξουμε την απαρτία. Χρειαζόμαστε, νομίζω, αν ήμασταν από την αρχή 12 ή 13 ε, στην αίθουσα. Έχουμε ήδη απαρτία με 11, δεν χρειάζεται και τους remote συμμετέχοντες. Θα ψηφίσουμε για το σύστημα ιδίων πόρων λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα EU for Health, το React, EU και τον μηχανισμό, ε, τον ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Κυρίσω την έναρξη της προφορίας τώρα έως τις ε, 5 παρατέταρτο, 16 και 45. Λίγη τώρα η συνεδρίασή μα και θα συναντηθούμε και μετά για την ανταλλαγή απόψεων με, με τον ε, Γερμανό Υπουργό, τον κύριο Ροτ, όχι σε αυτή την αίθουσα, στο 2Q2. 2Q2. Ευχαριστώ. <laughs> I saw you. <laughs> I was so concentrated. <laughs>